Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου δυστυχώς ο μιλητής. Κύριε Μπούντα, μικρόφωνο. Συνάδελφοι, οι εποχιακά εργαζόμενοι και οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι είναι απαραίτητη κατηγορία για πολλούς τομείς της οικονομίας και με τη, την κρίση του κορονοϊού διαπιστώσαμε ε, ότι η έλλειψή τους ε, θέτει σε κίνδυνο και την ύπαρξη ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Βρεθήκαμε λοιπόν βρεθήκαν σε πολύ δύσκολη ε, θέση και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει μηχανισμούς ώστε να μπορεί να διασφαλίσει ε, ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες για τους ανθρώπους αυτούς. Όσον αφορά τον τόπο όπου μένουν, τη διαμονή τους, ε, θα πρέπει να ε, ε, είναι επαρκής, θα πρέπει να έχουν επαρκή ιατρική ασφάλιση, για παράδειγμα. Επίσης, θα πρέπει να είναι δυνατό να ασκούν τα δικαιώματά τους και να μην αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μπούτα η κυρία Τούρα Φεράντης. Ε, Σας ευχαριστώ. Η πανδημία αποκάλυψε ότι η κινητικότητα των μεταναστών εργαζομένων στην Ευρώπη δεν σέβεται πάντα την ισότιμη μεταχείριση με τους υπηκόους της χώρας αυτής και Μιλώ και για τους ε, Ευρωπαίου υπηκόου αλλά και τους υπηκόου τρίτων χωρών όπως ισχύει για του εποχιακούς εργαζομένους στη Γεωργία που τόσο συνέβαλαν στον επιστημιστικό ανεφοδιασμό κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είδαμε περιπτώσεις ε, ε, επισφαλών, ιδιαίτερα επισφαλών συνθηκών ε, και επικίνδυνων για την υγεία και την προστασία τους. Επίσης, ε, εντοπίσαμε και απάτες και καταχρήσεις, γιατί είναι βάροτες αυτές οι ομάδες και αυτές οι καταχρήσεις δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό και πλήττουν την εικόνα του κλάδου. Επίσης, συμβαίνει και σε άλλους τομείς, στους οποίους υπάρχουν κάποια απαταιώνες μεσάζοντες που προσπαθούν να ε, στρατολογήσουν εργαζομένους στη μία χώρα και να τους μεταφέρουν σε άλλη για να εργαστούν σε άθλιες συνθήκες, όπως συνέβη με Ισπανούς, ε, Βούλγαρους και Ρουμάνους εργαζόμενους στις κάτω χώρες. Είναι απαράδεκτο σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει όλοι ε, χωρίς εξαιρέσεις να έχουν αξιότι, αξιόλογες και αξιοπρεπείς συνθήκες ασφαλείας εργασίας διαβίωσης άσχετα με τη χώρα πρόέλευση ή προορισμού του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Η συνάδελφος Κλεμπνή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία σύνταξη του ψηφίσματο αυτού για του διασυνοριακού και εποχιακού εργαζομένου στα πλαίσια τη πανδημία COVID-19. Σίγουρα δεν μάθαμε τώρα την κατάσταση, απλώ με την κρίση διευρύνθηκε. Σίγουρα είναι θεμελιώδης δικαίωμα αυτό των εργαζομένων και θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Δυστυχώ, η πανδημία έδειξε τις μεγάλες καταχρήσει και παραβιάσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που κανονικά θα πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη. Επιμένουμε λοιπόν στην ανάγκη να εξασφαλιστεί στου διασυνοριακού και εποχιακού εργαζομένου κατάλληλη κοινωνική προστασία και κατάλληλε εργασιακές συνθήκε και συνθήκε υγιεινής και προστασία. Επίση, έχουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία, τις επιθεωρήσεις εργασία. Θα πρέπει στα κράτη-μέλη το συντομότερο δυνατόν να εφαρμόσουν την αναθεωρημένη οδηγία για του αποσπασμένου εργαζόμενου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Συνήθως δεν δίνω τον λόγο ε, στους συναδέρφους που δεν ήταν παρόντες. Ε, ο κύριος Αντασόφσκι όμως καθόταν σε, σε άλλη θέση. Μάλλον, ποια είναι η θέση του. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Συνάδελφοι, Συμφωνώ με την πρόταση ψηφίσματος για τους διασυνοριακούς και εποχιακούς εργαζομένους. Είναι γνωστό ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι προέρχονται συνήθως από τις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες, ε, προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή τρίτες χώρες. Οι συμβάσει εργασία τους είναι ε, χρονικά περιορισμένες, οι συνθήκες εργασίας τους ε, είναι πολύ κακές. Συχνά ε, εργάζονται με αμοιβή χαμηλότερη από τον βασικό μισθό. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας αυτών των εργαζομένων. θα πρέπει οι συνθήκες υπό τις οποίες ε, εργάζονται να ε, συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Φανταστείτε Γάλλοι, Σουηδοί να πρέπει ε, να εργαστούν κάποια μέρα στην Ανατολική Ευρώπη και υπό τις ίδιες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό ο κύριος Ράιλ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, στην Γερμανία έχουμε ε, ένα νέο ξέσπασμα του κορονοϊού ε, στην κρεατοβιομηχανία και οι εργαζόμενοι αυτοί προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και τι λέει ε, ο Πρωθυπουργό τη Βόρεια Ελληνανία ε, Βεσφαλία, λέει ότι δεν φταίνε ε, οι συνθήκε διαβίωση και εργασία των ανθρώπων αυτών που μοιάζουν με σκλαβιά. Λέει ότι φταίει ότι πηγαίνουν στο σπίτι του, πηγαίνουν στην πατρίδα του το Σαββατοκύριακο. Με εκπλήσει πάρα πολύ ε, μια τέτοια δήλωση. Ε, ε, να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους αυτούς επειδή πήγανε στην πατρίδα τους και ότι γι' αυτό μας κολλάνε, αυτό νομίζω ότι είναι ξενοφοβική δήλωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νάιντκε, παρακαλώ κατώνες περιπτώσεις κορονοϊού σε σφαγείο στο Γκίτερσλο. και το ότι ο Πρωθυπουργό τη Βόρεια Γερμανία Ασφαλεία λέει ότι οι Ρουμάνοι ε, ε, ε, εργαζόμενοι φέρνουν αυτή την ασθένεια είναι απαράδεκτη, διότι έτσι ε, αρνείται τη δική του ευθύνη, διότι οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι εργαζόμενοι είναι ευθύνη επίσης ε, του Πρωθυπουργού της ε, Βορειά Γερμανία Βεσφαλία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε Πρωθυπουργό που να προστατεύει τους εργαζομένους ε, ασχέτως της εθνικότητάς τους και έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εργασίας ε, που να επιβλέπει την εφαρμογή των κανόνων. Θα πρέπει να δώσουμε τέλος σε τέτοιου είδους εκμετάλλευση ανθρώπων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράιντ. Αγγιλάρ, ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου αναγνωρίζοντα το τεράστιο έργο των εποχιακών εργαζομένων στη Γεωργία. Η κρίση μα θύμισε πόσο μεγάλη σημασία έχουν. Με βάση τι γεωργικέ οργανώσει ε, στην Ισπανία, δεν ε, μπόρεσε να γίνει εισοδεία ε, φρούτων λόγω τη πανδημία και 100.000 θέσει απασχόληση έμειναν κενέ. Γι' αυτό αγανακτώ που ένα τμήμα της κομμουνιστικής κυβέρνησης της χώρας ε, με παραπληροφόρηση κατηγορεί για όρους κλαβιάς τους ε, Ισπανούς γεωργούς, κάτι που πλήττει την εικόνα της ε, Ισπανικής γεωργίας ενός στρατηγικού κλάδου ιδιαίτερα όταν είδαμε πόσο έμειναν μερικές φορές άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιες κατηγορίες, πόσο χάναν τη ζωή του 40.000 Ισπανοί, 20.000 μάλιστα σε γυροκομεία χωρίς καμία οικονομι... Ε, υποστήριξη. Ε, στερήθηκαν οι Ισπανοί τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας. Ε, το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να ζητά συγγνώμη και όχι να κατηγορεί ε, τον Ισπανικό λαό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο κυρία με έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα μέτρα που έχουν λάβει τα κρατη και για την καταπολέμηση του ιού οδήγησαν σε καθεστώς ε, δυσχερών συνθήκων για του ε, διαστοριακού και εποχιακού εργαζόμενου και κυρίω σε εργαζόμενου ε, που εργάζονται στον κλάδο τη γεωργία χωρί ε, στέγαση, χωρί μεταφορά, χωρί προστασία τη υγεία του ζουν αυτοί οι άνθρωποι και θα ήθελα να μιλήσω για του εποχιακού εργαζόμενους συγκεκριμένα στον αγροτικό κλάδο οι οποίοι πραγματικά είναι αντικείμενο του καταχρα... εκμεταλλεύονται. Και αυτό στην Νότιο Ιταλία αποτελεί μια σαφή απάντηση. Η απάντηση είναι πολύ σαφή, μάλλον σε ό,τι αφορά του εργαζόμενου αυτού. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Να ζητήσω, μάλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εγγυηθεί τα δικαιώματα όλων αυτών των εργαζομένων που δέχονται διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει στο Συμβούλιο να διατεθούν οι πόροι εκείνοι που χρειάζονται για την υποστήριξη των ανθρώπων αυτών και να μπορέσουν να υποστηρίξουν και τι επιχειρήσει με τη σειρά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γκέμα και τώρα ο κύριο Φούλα. Έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε επίτροπε το είπατε κι εσεί προηγουμένω η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή τη ευρωπαϊκή ένωση. όταν μιλάμε για εποχιακού εργάτε ή εργαζομένου που διασταυρώνουν σύνορα για να πάνε στην εργασία του μιλάμε για ανθρώπου για ανθρώπου με οικογένειε και ανάγκε που εξαρτώνται από το μισθό του. Ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν με την προσδοκία ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρώπη θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τους προφυλάξουμε. ο ρόλος ο δικός μας εδώ σήμερα είναι να τους δώσουμε το μήνυμα ότι κατανοούμε τις ανάγκες τους φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε τις εργασίες τους να τους προστατεύσουμε και ότι στεκόμαστε δίπλα τους και όχι απέναντί τους. αυτό το μήνυμα πρέπει να φύγει σήμερα από αυτή την αίθουσα. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φουρλά. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Σαντζέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, η κρίση του COVID-19 αποκάλυψε ένα διαθετικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε τι γίνεται με τους εργαζόμενους και καλό και τους και τους εργοδότες μάλλον και τις ε, χώρες μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά τους εποχιακούς εργαζομένους. Από πλευρά ε, των κρατών μελών βλέπουμε ότι η λιτότητα έχει καταλήξει το καθεστώς πρόνοιας και τελικά ε, η Ευρώπη έχει αποτύχει. Πολλέ είναι οι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ε, δημοσιεύτηκαν, αλλά τι συνέχεια δόθηκε σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες αυτέ γραμμές. Εμείς οι σοσιαλιστές ζητούμε λοιπόν πιο πολύ διαφάνεια και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να αναλύει τον αντίκτυπο των μέτρων που ε, υπήρξε λόγω του κλεισίματο των συνόρων και ελπίζουμε η τα συμπεράσματα αυτά να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την νομοθετική πρόταση που θα κατατεθεί. Και εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να ευχαριστήσω τι πολυάριθμε ε, ΜΚΟ και του ε, κοινωνικού εταίρου που βοήθησαν σε αυτή την περίοδο κρίση του εργαζομένου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Πίλτα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πανδημία COVID-19, όπως ξέρετε, έπληξε βαρύτατα την οικονομία της Ευρώπης και στα πλαίσια αυτού του γενικού μαρασμού λαμβάνω το λόγο για να προασπίσω την νεολαία μας. Σε μια χώρα σαν τη Γαλλία που προβλέπει ένα εκατομμύριο ε, ανέργους, οι φοιτητές και οι νέοι πτυχιούχοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα οι νέοι θα βρουν θερινέ θέσει απασχόληση για να μπορέσουν να επιβιώσουν τον υπόλοιπο χρόνο, οι φοιτητέ δεν θα βρουν στάζ για να επικυρώσουν τα διπλώματά του, οι νέοι απόφοιτοι και πτυχιούχοι ε, θα ψάχνουν για μήνες ή για χρόνια μια θέση απασχόλησης στον τομέα των σπουδών τους. οι νέοι ονειρεύονται να φύγουν από την Ευρώπη για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Και κατά τη διάρκεια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει να σεβαστούμε τα, τους πιο αυστηρούς κανόνες ε, του, της εμποροκρατίας και να αφήσουμε στις χώρες μας να εισρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες αποσπασμένοι εργαζόμενοι και να μην δώσουμε ε, προτεραιότητα στη δική μας απασχόληση. Πριν μας ε, επιβάλλει το απαράδεκτο της δόγμα Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να σκεφτούμε τους νέους μας, τους αποφύτους μας, τους φοιτητέ μας, γιατί αυτοί θα γράψουν την... Δυστυχώς διακόπτεται το μικρόφωνο από τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Επόμενος ο κύριος Άνδρες έχει το λόγο. 55 χρονών περίπου, ήταν από τη Ρουμανία, ε, κατέρευσε ε, στην, ε, πάνω στην παραγωγή. Οι συνάδελφοί του έβριζαν γι' αυτό, έπρεπε να συρθεί χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει σπίτι του για να βρει έναν γιατρό. Εδώ στη Γερμανία κανένας δεν τον υποστήριξε. Έχουμε χιλιάδες διασνοριακούς εργαζομένους στα ναυπηγεία, στην καθαριότητα, στα σφαγεία. Πολλοί πληρώνονται ελάχιστα, ε, δεν έχουν καμία ε, ασφάλεια. Και ε, η κοινωνία ασχολείται με αυτούς μόνο όταν υπάρξει ξέσπασμα κοροναϊού σε σφαγεία. Δεν μας ενδιαφέρει ότι εκμεταλλευόμαστε τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει επιτέλους να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στον τομέα αυτών. Είναι θετικό ότι το Κοινοβούλιο με το ψήφισμα αυτό κάνει μια αρχή ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αντρέσεν. Η κυρία Σαλέψκα, ένα λεπτό. Panie Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πανδημία επιδίνωσε με τραγικό τρόπο ε, κάτι που είχαμε διαπιστώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Φυσικά αλλάζει συστηματικά η κατάσταση, αλλά εκεί που ήταν ήδη κακή έγινε πολύ χειρότερη. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να κάνουμε μια διεξοδική ανάλυση, να αντλήσουμε κάποια διδάγματα και να κάνουμε και κάποιες συστάσεις. Εμείς οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να επομιστούμε το καθήκον ε, και να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους από τις πατρίδες μας, γιατί οι συνάδελφοι στις Εθνικές Βουλές ε, είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των επιχειρήσεων που δεν ασφαλίζουν επαρκώς τους εργαζομένους και θα πρέπει από κοινού να λύσουμε τα προβλήματα. Η Γερμανική Προεδρία ελπίζω να έχει στο πρόγραμμά της και τέτοιου είδους ε, συζητήσεις με το, τους υπουργούς ώστε να μας παρουσιάσει μία έκθεση ε, και να προβληματιστούμε για όλα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό και να κάνουμε μία διεξοδική ανάλυση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γαλέσκα. Ο κύριος Πάλκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήμουν 16 χρονών όταν πέρασα κάτι εξετάσεις στο σχολείο μου και τότε οι γονείς μου ε, θέλησαν να μου κάνουν δώρο ένα ποδήλατο, αλλά χρειάστηκε να εργαστώ 21 μέρες ως ε, εποχιακά εργαζόμενος. Αλλά εργάστηκα με μεγάλη χαρά, μόνο το ποδήλατο μου σκεφτόμουν, χωρίς να σκέφτομαι την προστασία, την εργασία και την υγεία μου. Σήμερα βλέπω τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Γνωρίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκατομμύρια εποχιακοί και διασυναριακοί εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εγγυημένα δικαιώματα και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Ε, να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ασφάλειας, προστασίας και συνθήκες διαβίωσης. Η ευθύνη των εργοδοτών και των γραφείων πρόσληψης θα πρέπει να είναι αυξημένε. θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα εργασιακά τους δικαιώματα. Ευχαριστώ ε, του συντάκτες του ψηφίσματος γιατί έλαβαν υπόψη και τις δικές μας προτάσεις ε, του Ρουμανικού ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φάλικα. Μάγιο είναι ένα λεπτό. η πανδημία είχε τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή μας. Οι συνθήκες διαβίωσης και οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες ήδη ήταν στα όρια, μα πλήχθησαν πιο έντονα. Παρά το γεγονός ότι ήταν απαραίτητη η εργασία των ανθρώπων αυτών και χιλιάδες λοιπόν μετανάστες εποχιακά εργαζόμενοι, διεθνωρικοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στις, ε, στον τομέα της γεωργίας ε, εργάζονται υποφρικτές συνθήκες, χωρίς ρυθμισμένο ωράριο για ελάχιστους μισθούς και δεν ε, εγγυάται κανείς τις συνθήκες ε, εργασίας τους σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγεία. Τους εκμεταλλεύονται, τους εκμεταλλεύονται στην Ιταλία. Χρειαζόμαστε όμως και σχετικά μέτρα τα οποία θα επιβάλλουν την ίση μεταχείριση των εργαζομένων αυτών. Χρειάζεται λοιπόν να αντιληφθούν αυτές οι κοινωτικέ διατάξεις και για τους εποχιακούς εργαζόμενους και χρειάζεται φυσικά και σωστός προστατευτικός εξοπλισμός και για το πώς εργάζονται και δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί σε ό,τι αφορά τα ε, συμβόλαια εργασίας τους. Θα πρέπει να εγγυηθούμε το σωστό τρόπο εργασία του, να κινηθούμε κατά του κοινωνικού ντάμπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγιορίνο. Και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Κόντε. Θα πρέπει να ακούσουμε, να ακούσουμε όλους εκείνους που φτάνουν ε, στους εργαζόμενους, εποχιακούς και συναριακούς, με τις προσπάθειες να νομιμοποιήσουν τους παράτυπους εργαζομένους. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε πραγματικά στις ανάγκες εργατικών χεριών στις παραγωγικές μας δραστηριότητε, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους ε, χιλιάδες ε, συμπολίτε μας που έμειναν άνεργοι λόγω της κρίσης. Ακόμα και να εξετάσουμε το θέμα της έκδοση κουπονιών για, για προσωρινές θέσεις, για να μειώσουμε το φορολογικό άχθος. Επίσης, έχουμε κάποιους συμπολίτε μας που εξαρτούν τα έσοδά τους ε, στην εποχιακή εργασία. Για παράδειγμα, στα θέρετρα, οι εκπαιδευτές του σκι, οι ναυαγοσώστες, ε, οι ε, καθαρίστες, το προσωπικό καθαρισμού, οι σερβιτόροι στις, στα θέρετρα. Θα πρέπει να του εξασφαλίσουμε κατάλληλε και αξιοπρεπεί θέσει Μόνο έτσι θα έχουμε συγκεκριμένη προοπτική για να ξεφύγουμε από την κρίση. Σα ευχαριστώ. Με κύριο Σαγκάρτσε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η κρίση με το COVID-19 είχε σημαντικές επιπτώσεις ε, για τους δυσνοριακούς ε, εργαζόμενους και εγώ ζω σε μια περιοχή όπου ε, ισχύουν δίθες διατάξεις για αυτούς τους παίρνουν τα σύνορα. Είμαι σε, από ένα μέρος όπου είμαστε πολύ κοντά στο νεκρό αυτό κομμάτι και διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται η συνεργασία των κρατών μελών αυτών για να υπάρχει δυνατότητα μετακίνηση. Το ζήσαμε λοιπόν ιδιαίτερα στο, στην περιοχή μα το πρόβλημα και βλέπουμε ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα σαφέ μήνυμα προ του μετακινούμενου αυτού εργαζομένου, του εποχιακού εργαζόμενου, να στείλουμε από κοινού ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά την αξία τους, να αναγνωρίσουμε την αξία τους, γιατί πολλοί άνθρωποι φοβόντουσαν, ότι θα κλείσουν τα σύνορα και δεν ήξεραν πού θα μείνουν ε, τον επόμενο διάστημα, τον επόμενο μήνα, στο χώρο εργασία ή κοντά στην οικογένειά τους και χαρήκαμε που δόθηκαν, ε, δόθηκε βοήθεια και που στέλνει σαφές μήνυμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίγκρεσκου τώρα για ένα λεπτό. Συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα κοινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικό βήμα προόδου για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασία στου εποχιακού εργαζομένου. Είναι ένα ξεκάθαρο και χειρό μήνυμα. Δεν δεχόμαστε σύγχρονε μορφέ δουλεία. Εμεί οι σοσιαλδημοκράτε έχουμε ήδη ε, συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα και οι καταχρήσει που γίνονται στο εργατικό δίκαιο και στα κοινωνικά δικαιώματα. Στη Ρουμανία μάλιστα τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία εκατοντάδων εργαζομένων και δεν εφαρμόστηκε η ενωσιακή νομοθεσία. Το ψήφισμα ουσιαστικά επαναλαμβάνει κάτι που επανειλημμένως καταγγείλαμε στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και πάνω από 50.000 άνθρωποι υπέγραψαν τη σχετική μας ε, αναφορά. Φυσικά δεν θα είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα. Πολλοί προσέφηκαν στη δικαιοσύνη, αλλά όσοι συνοστίζονται στα φορτηγά και τι δαλίκε περιμένουν πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους που παραβιάζονται καθημερινά, όπω τα δικαιώματα των Ρουμάνων εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε στην Νιγκρέσκο. και τώρα το λόγο έχει η συνάδελφο για λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητάμε σήμερα εδώ το θέμα των εποχιακών εργαζομένων σε ό,τι αφορά το πλαίσιο τη ε, κρίση ε, COVID-19 και το θέμα είναι πώ θα χειριζόμαστε και τα σύνορα. Αυτά που συνέβησαν στην Ιταλία κατά τη διάρκεια τη κρίση ε, COVID-19 ήταν χιλιάδε οι παράνομοι εργαζόμενοι που έφτασαν στα σύνορά μα. Δεν λειτουργήσε λοιπόν σωστά η σύνορια φλέκη και σε ό,τι αφορά το θέμα τη καραντίνας, για παράδειγμα υπήρχαν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Βρέθηκαν ε, λύσεις ε, ad hoc για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά κανείς ε, δεν βοήθησε. Τι έκαναν λοιπόν οι κυβερνήσει δεδομένη τη ε, κριση covid COVID-19 δημιούργησαν ε, εξαιρέσει ε, για του εποχιακού εργαζόμενου. Παράλληλα όμω δεν είχαν δουλειά και εκατομμύρια Ιταλοί. Αυτό ήταν πραγματικά αποτυχία και τη Ευρώπη και τη Ιταλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνάδελφο κυρία Σαρντόνα. Ο κύριο Λούτσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση COVID έδειξε πόσο σημαντική είναι η εποχιακά εργαζόμενη για να καλυφθούν οι επιστηστικές ανάγκες ε, του συνόλου των Ευρωπαίων. Και σίγουρα οι εργαζόμενοι αυτοί χρήζουν ε, σεβασμού και της αναγνώρισης μας. Και ευχαριστώ το ψήφισμα που το αναγνωρίζει και βαίνει προς σωστή κατεύθυνση της προστασίας τους. γιατί είναι θεμελιώδης ε, πυλώνας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Επίσης υπάρχει και το θέμα των διασυνοριακών εργαζομένων. Ε, ειδικά στην πατρίδα μου έχουμε πολλούς. Θα πρέπει να τους διευκολύνουμε, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης. Είχαμε πολλές δυσκολίες στα σύνορα. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα είδος ε, διαβατηρίου εργασίας για τους διασυνοριακά εργαζομένους, για να διευκολύνουμε τους ελέγχους και να διευκολύνουμε και τις επιχειρήσεις που χρειάστηκε να καταφύγουν σε πολλές διοικητικές διατυπώσεις. Γιατί λοιπόν να μην οργανώσουμε κάτι τέτοιο σε διάφορα επίπεδα, εκδίδοντας ένα διαβατήριο πέντε αστέρων, για παράδειγμα, για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που χρειάζεται να περάσουν τα σύνορα για να παράσχουν υπηρεσίες υγείας στις παραμεθόριες περιοχές. Έτσι θα βελτιώσουμε, νομίζω, τη ζωή πολλών συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κόχουτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ για το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη μίλησα στην Ολομέλεια για την ανάγκη της προάσπισης των δικαιωμάτων των διασυνοριακά εργαζομένων. Θα ψηφίσουμε στην Ολομέλη αυτή ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, τα δικαιώματα των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων. Επί τη ευκαιρία μου και εγώ τέτοιο εργαζόμενο για μία πενταετία περίπου και είναι ένα καλό βήμα, ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που θα πρέπει να ακολουθήσει όμω είναι αυτέ συγκεκριμένε δράσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τα κράτη-μέλη. Και νομοθετικέ και μη νομοθετικέ προτάσει και μέτρα χρειάζονται κυρίως η παροχή σημαντικών πληροφοριών και σωστή ενημέρωση. Γιατί δεν έγινε σωστή ενημέρωση στη διάρκεια της κρίσης. Δεν προστατεύσαμε τους διασυνοριακούς εργαζόμενους στη Εκκλησίας. Εγώ μόνος μου άνοιξα στο γραφείο μου ένα διασυνοριακό γραφείο επαφής γιατί το κράτος ήταν απόν. Λάθος είναι κάτι τέτοιο. Ε, οι κοινωνίες μα είναι ανθεκτικέ, ιδιαίτερα όταν είναι καλά ενημερωμένε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε επίκαιρες ε, και καλές πληροφορίες για τους διασυνοριακά και για εποχιακά εργαζομένους, γιατί είναι σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα κάτι τέτοιο. Ολοκληρώνονται λοιπόν έτσι οι εισηγήσει των αμελητών. Ε, ε, το λόγο έχει ο Επιτροπός Σμιτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, σήμερα συζητήσαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικοδομήματο, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Είναι ένα μεγάλο πλέον έκτημα μία μεγάλη επιτυχία, ένα μεγάλο επίτευγμα, αλλά συνεπάγεται και μεγάλες ευθύνε. Δυστυχώ. Υπό το φως της τρέχουσας κρίσης διαπιστώσαμε ότι κάναμε βήματα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά αυτή την ελευθερική κυκλοφορία υπάρχουν καταστάσεις απαράδεκτες, συνθήκες εργασία, οι οποίες δεν θεωρούνται αξιοπρεπεί, συνθήκε διαβίωσης οι οποίες είναι απαράδεκτες. Η συζήτηση λοιπόν αυτή θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε με πιο αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο τα προβλήματα αυτά. Δεν είναι μία λύση, όπως είπαν κάποιοι, να αφήσουμε κατά μέρος την οδηγία για την από το για τους αποσπασμένου, γιατί αν ε, είχε σωστά εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, δεν θα ήταν ε, η κατάσταση όπως είναι, ε. Και δεν είναι το πρόβλημα η ένομη κατάσταση, η νόμη. Το θέμα της υλοποίησής τους είναι που χωλαίνει. Η έλεγχη είναι αυτή που είναι ανεπαρκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση σε όλου και σε όλε, προφανώ και στου εργοδότε, προφανώ και στα κράτη-μέλη, να εφαρμόσουν σωστά την νομοθεσία, τι αρχέ, τι ευρωπαϊκέ. Και νομίζω ότι αν το πετύχουμε αυτό, θα μπορέσουμε να πετύχουμε πρόοδο και θα μπορέσουμε να επανακτήσουμε την αξιοπρέπεια που αξίζει σε όλου αυτού του εργαζόμενου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε Σμιτ. Και τώρα το λόγο έχει πάλι από το Συμβούλιο η Υπουργό Πρινιάτση. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Κλείνοντα, ε, θα ήθελα να επαναλάβω την υποστήριξη του Συμβουλίου ε, στην ελεύθερη μετακίνηση των ε, διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων. Θέλουμε να παράσχουμε στους εργαζόμενους αυτούς την ίδια μεταχείριση με τους εθνικούς εργαζομένους και μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητούμε την καλύτερη λύση για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που μας έφερε ο ιός. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ αν κατάλαβα σωστά. Αυτή είναι η τελευταία παρέμβασή σας ε, με την ιδιότητα ε, της Προεδρεύοντος ε, του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον και ελπίζω στο μέλλον να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Έληξε η συζήτηση, θα πραγματοποιηθεί αύριο η ψηφοφορία. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 6 και 4. Πού Ο κουπολεύει